Πρώτη εξέταση τη έκθεση ιδία πρωτοβουλία για, για την κατάσταση σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑ με τον κύριο Μπρόκ ω εισηγητή. Θέλετε να συνεχίσετε, κύριε Μπρόκ. Δική σα είναι η έκθεση. Βλέπω ότι δεν υπάρχει διαφορά στο ακροατήριο, οπότε θα παραμένω στα προηγούμενα σχόλιά μου. και ευχαρίστως να ακούσω τις παρατηρήσεις ε, των συναδέλφων εκεί που ενδεχομένως να χρειαστεί αναδιατύπωση, διόρθωση. Θα ήθελα τις απόψεις των ε, συναδέλφων και τις προτάσεις τους. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόκ. Το σχέδιο της έκθεσης στα αγγλικά σας έχει αποσταλεί με mail, οπότε διατέθηκε σε όλες τις γλώσσες κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Πρέπει να ακούσουμε τους σκιώδεις πρώτα για ε, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Πάσκου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποστινάρο είναι στην πραγματικότητα ο σκιώδης εισηγητής, αλλά δυστυχώς δεν είναι στις Βρυξέλλες. Επέστρεψε στη Ρουμανία για ιατρικό του θέμα και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Οπότε αναγκαστικά θα διαβάσω τα, ε, αυτά τα ολίγα που μου έχει ε, εγχειρήσει και στα αγγλικά για να το ευχαριστηθούν όλοι. Ιδίως ο Χέλμουτ. Αφού απαριθμώνται οι παράγοντες που κάνουν τις διατλαντικές σχέσεις να είναι τόσο σημαντικές όσο ήταν πάντοτε, Ο κύριος Μποστινάρου πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στην έκθεση. Αρχίζω λοιπόν να διαβάζω. Φοβάμαι ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε, να αναγνωρίσουμε και κάποια λάθη του παρελθόντος, ε, όπως η παρέμβαση στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και το πόσο αποσταθεροποίησαν ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα πρέπει να έχει πιο δραστηριό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία ε, λύση ειρήνευσης ε, μακροπρόθεσμη για τη Μέση Ανατολή και για να προστατεύσουμε τη Συμφωνία των Πυρηνικών με το Ιράν αναζητώντας διπλωματική επίλυση στο θέμα της εμπλοκής του Ιράν στην σύγκρουση της ε, Συρίας. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα απαραίτητο, το απαραίτητο πρόγραμμα για την ε, σταθεροποίηση της κατάστασης στην Συρία. Θα πρέπει μέσω της ανατολικής Γετονίας να δούμε σοβαρά την παρουσία της Ρωσίας στην ε, Συρία και την, και την όλη της εμπλοκή η έκθεση αυτή πρέπει να είναι σαφέστερη και να επικεντρώνεται σε αυτές τις προτεραιότητες καθώς και την ενίσχυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του ΟΗΕ, ζητώντας καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει ένα ενιαίο μέτωπο. Και από την επιστολή του συναδέλφου, και μια δική μου παρατήρηση πέρα από όσα διάβασα. Για μένα, στον κόσμο μας σήμερα, ούτε και οι ΙΠΑ δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνες τους. Αργά ή γρήγορα θα χρειαστούν συμμάχους. Γι' αυτό να έχουμε υπόψη ότι είναι λίγο παράτολμο να λέμε δεν μπορώ να, να, ότι δεν χρειάζομαι κανένα και μπορώ να τα καταφέρω όλα μόνο μου. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Ευχαριστούμε κύριε Πάσκου. Επειδή δεν βλέπω να είναι εδώ όλοι οι συγητέ. Θέλει κάποιο άλλο από του σκιώδε το λόγο. Από του σκιώδε πρώτα. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μιγιανμόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο. Δυστυχώ την έκθεση του κυρίου Μπρόκ δεν είχα χρόνο να τη διαβάσω. Την έλαβα μόλι σήμερα και μάλιστα το απόγευμα. Πάντω, επειδή έχω υπάρξει εγώ ίδιο εισηγητή στο παρελθόν για τέτοιου είδου σχέσει, είπα και Ευρωπαϊκή Ένωση επί Ομπάμα, αυτό που μπορώ να κάνω καταρχάς είναι να ευχαριστήσω τον κύριο Μπροκ για τις προσπάθειές του, διότι τουλάχιστον αναφέρεται στα βασικά σημεία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα η έκθεση του κύριου Μπροκ, ασχέτως του ποιος έχει αναλάβει καθήκοντα στο Λευκό Οίκο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ καλό και οι αρχικές ε, παράγραφοι επικεντρώνονται στη στατική σχέση, η οποία ελπίζουμε ότι δεν θα αλλάξει παρά τις ε, ταραχώδες στιγμές που τώρα ζούμε. Στην προηγούμενη συζήτηση είδαμε να λέγεται ότι τα πάντα τελειώνουν κάποτε, αλλά έχουμε πολλές δεκαετίες πίσω μας κοινών συμφερόντων, κοινών επιδιώξεων, κοινών αξιών. Αυτό ελπίζουμε ότι θα εξακολουθήσει. Και είμαστε ανέκαθεν σοβαροί σύμμαχοι και εταίροι για τους δε. Αυτό σωστά τονίζεται στο κείμενο και τον ευχαριστώ τον κύριο Μπροκ, καθώς και για το ότι συμπεριέλαβε την ιδέα να υπάρξει ένα διατλαντικό πολιτικό συμβούλιο, κάτι που έχει ακουστεί και στο παρελθόν ως ιδέα. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και θα χαιρόμουν να έβλεπα να γίνει πραγματικότητα η πρόταση του κυρίου Μπροκ. Ο κύριος Μπροκ συμπεριέλαβε σωστά την ιδέα αυτή στο σχέδιο έκθεσης. Βεβαίως, θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο για να μελετήσω το σχέδιο έκθεσης με προσοχή, αλλά Στην παράγραφο για τι διμερεί σχέσει, εκεί που γίνεται λόγο για την ενίσχυση τη στρατηγική μα εταιρική σχέση, πρέπει τα μηνύματα μα να είναι εμπορικά αλλά και οικονομικά. Δηλαδή να υπογραμμίσουμε και τη διάσταση του κέρδους. Βεβαίω θέλουμε να συσφίξουμε τους οικονομικούς δεσμούς, τους εμπορικούς δεσμούς, όμως ε, εδώ ε, αυτό που είναι ρεχοκοκαλιά αυτών των σχέσεων είναι το χρήμα και πρέπει να αναζητήσουμε και την κατάλληλη διατύπωση. Σε κάθε περίπτωση εδώ δεν έβαλε στον πάγο την Συμφωνία ΔΕΤΗΠΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό που θέλουμε είναι μια αμοιβαίω φιλόδοξη εμπορική συμφωνία. Όχι απλώ να ασχολούμαστε με εμπορικά μέτρα, αλλά να έχουμε μέτρα που εξασφαλίζουν πρόσβαση στι δημόσιε προμήθειες λόγου χάρη, όπω λέει ο κ. Γκάρτνερ. Στι παραγράφου λοιπόν 1 έω 12 καλό είναι να συμπεριληφθεί η ιδέα ότι θέλουμε εντονότερου εντονότερους οικονομικούς δεσμούς σε σχέση με αυτό που πιστεύει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Και δεν νομίζω ότι το τονίζουμε αρκετά ως τώρα. Αυτή είναι η μόνη ε, μικροπροστίκη που θα πρότεινα ε, και που θεωρώ ότι θα βοηθούσε αρκετά το κείμενο. Ευχαριστούμε κύριε Μιγιανμόν. Ζητά κανένα άλλο το λόγο. Εάν όχι, θα σας δώσω το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη εξέταση ήταν σήμερα, όπως καταλάβατε. Ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 7 Ιουνίου 11 το πρωί. Μετά έγκριση στην Επιτροπή ΙΝΤΑ της νομοδότησης ΙΝΤΑ 20 22 Ιουνίου. Εξέταση στην Επιτροπή μας 10-11 Ιουλίου. Ε, επίσης τον Ιούλιο στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Κύριε Μπροκ, έχετε τίποτα να σχολιάσετε. Εάν όχι, ολοκληρώνουμε με το σημείο αυτό. Α. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Μιλαν για την προσθήκη που πρότεινε ε, στην έκθεση. Ε, και κάποια άλλα σημεία της έκθεσης θα έχω πάρει από προηγούμενη δική του έκθεση, δεν θα πρέπει λοιπόν να επενεθώ εγώ γι' αυτά. Θα εξετάσω τις παρατηρήσεις που έγιναν. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροπολογιών. Έχουμε φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Ε, εργαζόμαστε με βάση έναν κοινό, κινούμενο στόχο. Θα, δούμε, θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Όταν θα έχουμε τις τροπολογίες ε, θα γίνει και σχετική συζήτηση. Θα πρέπει όμως να εργαστούμε ώστε να μην καταλήξουμε ε, με μια κακή έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόκ. Ελπίζουμε όλα να προχωρήσουν ομαλά. Έτσι ολοκληρώνουμε την ε, συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Σε τρία λεπτά θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα μας. Ανταλλαγή απόψεων με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, επικεφαλής της αποστολής Γιούλεξ Κωσυφοπαίδιο. Τρία λεπτά. Όπω είπα, έχουμε το σημείο 17 τώρα, ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, επικεφαλής της αποστολής Γιούλεξ Κωσυφοπέδιο. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσουμε την κυρία Παπαδοπούλου, επικεφαλής της αποστολής στήρησης του ε, δικαίου στο Κωσυφοπέδιο, τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία εννέα χρόνια η Γιούλεξ παρακολουθεί το κάτω δικαίου και τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις στο Κωσυφοπαίδιο, προσπαθώντας να ελέγξει την κατάσταση εκεί η νέα εντολή προς τη Γιούλεξ από τις 14 Ιουνίου μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες της Γιούλεξ για να παρακολουθήσει καλύτερα το τι συμβαίνει στην πράξη. Η κυρία Παπαδοπούλου προωθεί, ε, εργάζεται ε, για τα θέματα της διεύρυνσης και ε, που παραμένει μια στρατηγική προτεραιότητα για την Επιτροπή αυτή. Μιλάμε εδώ για έξι χώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το κοσυφοπαίδιο καθώς μας απασχολεί να υπάρχουν καλές σχέσεις γειτονία και το κράτος δικαίου. Βεβαίω εδώ ε, πρέπει να πούμε ότι βεβαίως είναι δύσκολη η δουλειά της αποστολής ε, Γιούλεξ και ότι χρειάζεται ε, η πραγματική τεχνική οικονομική αρρωγή προς το κοσφοπέδιο. Βεβαίω η διεύρυνση προ τα Δυτικά Βαλκάνια είναι συμφέρουσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε να, υπάρχει να υπάρχουν σωστέ δαπάνε για να αξιοποιείται το χρήμα των φορολογουμένων και να μην ε, υπάρχει σφάλμα στον προγραμματισμό για μετά το 2020. Σε καμία περίπτωση κακοδιαχείριση παρατυπία τα σταλία μπορεί να ε, γίνει ανεκτή. Οι ατασταλίε στη Γιούλεξ απασχολούν ιδιαίτερα στο Ευρωκοινοβούλιο και περιμένουμε να δούμε να υπάρχει πλήρης διερεύνηση. Κυρία Παπαδοπούλου, ενώ διαμορφώνεται και ελέγχεται τη διαδικασία ελέγχου, εδώ Πρέπει ε, να έχουμε μια καλή συζήτηση με τους ε, εισηγητές για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ιδίως τον εισηγητή μας ε, για το κοσυφοπαίδιο. Μαζί μας είναι και ο κύριος Κένεθ Ντίν, υπεύθυνο για την κοινωνία των πολιτών και τι αποστολέ για την προάσπιση τη κοινωνία των πολιτών σε σχετικέ αποστολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν σα δώσω το λόγο, κυρία Παπαδοπούλου, να δώσω το λόγο στον κύριο Κένεθ Ντίν για να σα παρουσιάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα ευγενικά σα λόγια και την ίδια μα την αποστολή. Απλώ ήθελα να δώσω ένα-δύο στοιχεία σε σχέση με το περιεχόμενο και το τι έχει αναλαβεί η Αλεξάνδρα. Ε, η EULEX είναι τεράστια αποστολή από τότε που την συνέλαβαν οι δημιουργικές της και δείχνει πώς εξελίσσεται η κοινωνία των πολιτών στα πλαίσια της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ε, στα πλαίσια μιας αποστολής για το κράτος δικαίου. Ε, μιλάμε για μια θητεία, μια εντολή που στο κέντρο της είχε την ε, μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου στο Κωσυφοπαίδιο. Είναι μια δύσκολη αποστολή αυτή στο Κοσφοπέδιο, πάντοτε ήταν, αλλά δεν είχε, αν δεν είχε προβλήματα δεν θα βρισκόμαστε εδώ. Αυτό που μπορεί να πει κανεί είναι ότι η αποστολή όλα αυτά τα χρόνια με χιλιάδε συναδελφού να εργάζονται παγκοσμίω έχει ξεπεράσει πολλές δυσκολίες και έχει να παρουσιάσει επιτυχίες και επιτεύγματα. Βεβαίω, το κακό είναι ότι οι κακέ ειδήσει ταξιδεύουν γρηγορότερα από τα θετικά επιτεύγματα. Πάντω, νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ η αποστολή αυτή γίνεται ε, σεβαστή και από τον κόσμο στο κοσφοπέδιο και εκτό. Και χθε μπορέσαμε να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά και στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ στο Ευρωκοινοβούλιο και φάνηκε από τη συζήτηση ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς ε, διαπιστώσεις, προβλέψεις μάλλον, για το τι θα συμβεί Μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά δεν μπορούμε ως αποστολή να προβλέψουμε πώς θα διαμορφωθεί το κοσυφοπαίδιο. Ούτε αν η παρουσία μας θα φέρει μια πραγματική διαφορά στην πράξη. Σίγουρα υπάρχει μια ευρωπαϊκή παρουσία και υπάρχει καλύτερη διασύνδεση με την ευρωπαϊκή οικογένεια, καθώς και με τους διεθνείς εταίρους της ΕΠΑ, τον ΟΗΕ και τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους σε αυτή την περιοχή, για τα τοπικά αυτά προγράμματα αλλά η αποστολή έχει όντως ένα σοβαρό ρόλο στο κοσυφοπαίδιο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε φυσικά όλα, αλλά τα κράτη-μέλη μας έχουν δώσει τις ε, ε, εντολές τους το καθένα για τη μελλοντική μας δουλειά και επιτέλους μια παρατήρηση για αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Η Αλεξάνδρα είναι επικεφαλής της αποστολής και ε, ασχολείται με το κατά πόσο τηρούμε αυτά τα οποία ε, έχουμε αναλάβει στην εντολή. Η Αλεξάνδρα νομίζω ότι είναι άξια επικεφαλής και τη γάνει κάθε σεβασμού και είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να της δώσω το λόγο ευχαριστώντας τη για όλη τη δουλειά που συνεχίζει να κάνει. Που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει. Σας ευχαριστούμε κύριε Κένετ για αυτά τα ευγενικά σας λόγια. Κυρία Παπαδοπούλου, χωρίς καθυστερήσεις να σας δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για το καλωσόρισμά σας. Και σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Σας ευχαριστώ όλους που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να σας παρουσιάσω την αποστολή μας. Είναι πολύ ε, κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε την αποστολή αυτή, το παρελθόν και το μέλλον της, διότι, όπως μόλις ανέφερε ε, η κυρία Πρόεδρο, τον Ιούνιο λίγη η παρούσα ε, εντολή και βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, διότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε μόνο προσαρμογή με βάση τα νούμερα, θα έχουμε πλήρη ανανέωση της αποστολής. Θα έχουμε νέα αποστολή, διότι θα επικεντρωθούμε σε άλλα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν. Θα επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα ζητήματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα θα έχουμε πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογή σε σχέση με πριν. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην κατάσταση. Η κατάσταση στο κοσυφοπαίδιο δεν είναι η ίδια με πριν 10 χρόνια. Ε, έχουν πετύχει πολλά οι Κωσοβάροι. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτά. Συνεχίζουν να υπάρχουν όμως και προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και στα οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί η αποστολή. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τις επιτυχίες και τις προκλήσεις, τα 28 κράτη-μέλη μαζί με τα θεσμικά όργανα έχουν προχωρήσει και προσπαθούν τώρα να διαμορφώσουν μια νέα μεταβατική αποστολή. Το Κόσοβο βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς για να ε, αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Πρωτού φτάσω στο μέλλον, θα ήθελα να αναφέρω κάποια από τα επιτεύγματα του παρελθόντος, διότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε από πού ξεκινήσαμε. Και θα προσπαθήσω να σας δώσω και κάποια στοιχεία και κατόπιν Μπορεί ο καθένας να σχηματίσει άποψη σχετικά με το αν αποτελεί επιτυχία η αποστολή ή όχι. Από εκτελεστικής πλευράς, ε, ε, πάνω από 500 ε, αποφάσεις σε ποινικέ υποθέσεις, διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα, πάνω από 100 αστικές υποθέσεις, και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ιδιοκτησίας, όπου είχαμε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ε, περιπτώσεις, υπόπτους που συμπεριλάμβαναν ε, πολλούς εξωματούχους υψηλού επίπεδου, βουλευτές κλπ. Ταυτόχρονα, οι δικαστικοί εμπειρογνώμονές μας ε, έχουν παρακολουθήσει την κατάσταση και έχουν παράσχει συμβουλές στους κοσοβάρους ομολόγους τους. Έτσι ε, μπόρεσαν να οικοδομηθούν πιο ανθεκτικοί ε, οργανισμοί ε, αντί να βασιστούμε σε μεμονωμένα προγράμματα. Επίσης, ερευνήσαμε 251 περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου. Έτσι, ουσιαστικά διερευνήσαμε όλα τα εγκλήματα πολέμου στο Κόσοβο. Είχαμε τις υποθέσεις UNMIC, 98 νέες έρευνες ξεκίνησε η αποστολή μας, εκ των οποίων η πρώτη ε, είχε να κάνει με βιασμούς ε, και εγκλήματα πολέμου. Ήδη από την ε, αρχή της αποστολής μας, πάνω από 2.400 υποθέσεις δόθηκαν στον Γενικό Ισαγγελέα του Κοσφοπεδίου στην εισαγγελία στην ε, Μητροβίτσα καθώς και στην κινητή μονάδα εισαγγελέων. Η αποστολή μας ε, συμμετείχε σε διάφορα στάδια της διαδικασίας σε πάνω από 1.300 υποθέσεις ε, που συμπεριλαμβάνουν πάνω από 210 εγκλήματα πολέμου, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οικονομικό έγκλημα και άλλα. Ήδη από την αρχή οι εισαγγελείς της Γιούλεξ κατάφεραν να πετύχουν αρκετές καταδίκες σε περιπτώσεις ε, οργανωμένου εγκλήματος. Πέρα από τον αριθμό των υποθέσεων με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί, ε, το εγκληματολογικό εργαστήριο έχει εκτελέσει ε, πάνω από 600 επιτόπου επιχειρήσεις ε, και έχει εξετάσει πάνω από 400 υποθέσεις. Επίσης έχει προσπαθήσει να εντοπίσει αγνοούμενους ε, Χιλιάδες έγγραφα εξετάστηκαν και 2.300 δείγματα οστών εστάλησαν για ταυτοποίηση. Επίσης έχουμε παράσχει νομοθετική βοήθεια στις αρχές ε, του κοσφοπεδίου. Ε, έχουμε ε, βοηθήσει στην διατύπωση πάνω από 150 νόμων. Επίσης έχουμε βοηθήσει στις οργανωτικές τροποποίησεις στα τελωνία του κοσφοπεδίου. Κάτι που έχει οδηγήσει σε ανάκτηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ε, από την έναρξη των επιχειρήσεών μας στο αεροδρόμιο της ε, Πρίστινα έχει ε, βελτιωθεί η ανάκτηση οικονομικών πόρων κατά πάνω από 500%. Επίσης, ο φορέας μας θεωρείται ένας από τους πιο αντικειμενικούς και σεβαστούς στο κοσυφοπαίδιο. Ε, έχουμε βοηθήσει και στην επάνδρωση ε, σημείων διέλευσης των συνόρων. Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τοπικές αρχές ε, για να στηρίξουμε την δημιουργία των έξι μόνιμων σημείων διέλευσης των συνόρων. ασχολούμαστε με την εφαρμογή της ε, Συμφωνίας ε, Ελεύθερης ε, Κυκλοφορίας και από τις 15 Νοεμβρίου 2014 οι σχετικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνουν και δύο αεροδρόμια. Έχουμε μία ομάδα έγκαιρης παρέμβασης Επίσης ε, στηρίζουμε την ε, ενσωμάτωση Κωσοβάρων ε, στην βόρεια μονάδα της αστυνομίας και 2,5 χιλιάδες βιβλία ληξιαρχικά που βρέθηκαν στην Σερβία έχουν παραδοθεί. Επίσης, προσχώρησαν στο δικαστικό σύστημα του Κωσόβου 40 δικαστές από τη Σερβία. Αυτά όσον αφορά το παρελθόν. Ας προχωρήσουμε τώρα στο μέλλον. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να αναφέρω ότι τα τελευταία 10 χρόνια 10.000 άνθρωποι έχουν εργαστεί στην Ιούλεξ και πρέπει να επισημάνουμε την συνεισφορά τους καθώς και η δουλειά όλων των προκατόχων μου που πέτυχαν τόσα πολλά υπό τόσο δύσκολες συνθήκες. Η νέα αποστολή θα πρέπει να εξετάσουμε την διαμόρφωση, τη διατύπωση της νέας έντολης. Ε, πρέπει να ασχοληθούμε με τη διαχείριση κρίσεων στο Κωσυφοπαίδιο. Το Κωσυφοπαίδιο τώρα πια ξεφεύγει από το στάδιο ε, διαχείρισης της κρίσης. Πρέπει λοιπόν τώρα να αναγνωρίσουμε τα επιτέματα του Κωσυφοπαίδιου και να προχωρήσουμε σε άλλες μορφές ε, βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει το Κωσυφοπαίδιο επειδή φεύγει η Ιούλεξ. Οι δραστηριότητε παρακολούθησής μας ε, θα αναλυθούν από άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συχνά με τη βοήθεια μεμονωμένων κρατών μελών και διεθνών εταίρων. Από τους ε, τρεις ε, τομείς όπου η Γιούλεξ είχε συμβουλευτικό και, ε, ρόλο και ρόλο παρατηρητή, η βοήθεια αυτή θα συνεχιστεί από άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι επιμέρους προγράμματα. Όσον αφορά την διαφθορά όπου πρέπει να γίνει ακόμη δουλειά, η παρακολούθηση και η παραχή συμβουλών θα συνεχίσει να παρέχεται από την Ιούλεξ. Είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να υπογραμμίσω την ε, εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, Πρίστινα. Ήταν πολύ σημαντικό για τις Βρυξέλλες ότι ήταν τόσο ομαλή η μετάβαση αυτή και στο πλαίσιο αυτό. Η στενή συνεργασία μας με άλλους φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε ευγνώμονες απέναντι στους συναδέλφους μας στην EUSR για την εξαιρετική συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ψηφοπαίδιο να καταλάβει ότι ε, πάρα πολύ σημαντικά στο μέλλον ε, θα είναι η δημιουργία δυναμικού και η σωστή συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό του στη διαδικασία αυτή, όχι απαραίτητα όμως υπό τη μορφή της Ιούλεξ. Η νέα ε, εντολή δίνει τέλος στον εκτελεστικό μας ρόλο. Από τις 14 ε, Ιουνίου του 2014 δεν θα υπάρχουν πια εισαγγελείς ε, στο δικαστικό σύστημα του Κωσοπεδίου. Πέρα όμως από τις υποθέσεις ε, που ήδη έχουν φτάσει στο δικαστήριο, υπάρχουν διάφοροι, διάφορα αρχεία τα οποία δεν μπορούν ακόμα να περάσουν στο δικαστήριο ή όπου τα στοιχεία είναι πενιχρά όλες αυτές οι υποθέσεις ε, θα πρέπει να διαβιβαστούν στις τοπικές αρχές. Η δουλειά αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και αποτελεί πολύπλοκο έργο, διότι μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες σελίδων που πρέπει να ε, μεταφραστούν στα αλβανικά και τα σερβικά και οι φάκελοι αυτοί θα πρέπει να αξιολογηθούν από την αστυνομία και τους εισαγγελείς και θα πρέπει να παραδοθούν με πολύ συντεταγμένο τρόπο, διότι η Γιούλεξ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις υποθέσεις αυτές και να παρέχει συμβουλές και βοήθεια στους ε, Κωσοβάρους ομολόγους μας, διότι είναι πράγματι ε, τεράστιο το έργο αυτό. Η Γιούλεξ με τη νέα εντολή της ε, θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια και είναι αυτονόητο ότι ο ρόλος μας είναι να ε, στηρίξουμε την Χάγη. Βέβαια δεν ήταν ε, όλα τέλεια ήδη από την αρχή. Επρόκειτο για την ε, πρώτη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκτελεστική εντολή σε μια περιοχή με πολύ αστάθεια. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν άδικο να περί κανείς ε, ότι όλα θα πήγαιναν τέλεια. Το μεγαλύτερο λάθος πιθανότατα ή έπασε το ο τομέας όπου θα έπρεπε να έχουμε χειριστεί τα πράγματα διαφορετικά ε, ήταν η διαχείριση των προσδοκιών των Κωσοβάρων, των κρατών μελών και ακόμη και των δικών μας προσδοκιών. Έχουμε ένα χώρο με πολλά προβλήματα στο κράτος δικαίου. Ένα χώρο που, μια χώρα που ξέφυγε από μια εμπόλεμη σύγκρουση. Πετύχαμε όσα μπορούσαμε και νομίζω ότι ως Γιούλεξ, Γιούλεξ κάναμε περισσότερα από ό,τι περιμέναμε, αν και πρέπει να γίνουν και άλλες βελτιώσεις. Πολλοί αναρωτιούνται πώς βοηθάει το κοσυφοπαίδιο η Ulex. Βεβαίως είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς αυτή την ερώτηση, γιατί παρόλο που η Γιούλεξ ε, επί χάρτου είναι μια τεχνική αποστολή, δεν μπορούμε να ε, υποτιμούμε τις πολιτικές συνέπειες τη δουλειά τη. Υπ' αυτήν την έννοια η Ulex είναι μέρος του πολιτικού συστήματο στο κοσυφοπαίδιο ακόμη και εμέσω. Μέρος του πολιτικού σκηνικού, ιδίω στο κοσυφοπαίδιο, αντιμάχεται τη Γιούλεξ. Για να το πω απλά, κάποιοι περίμεναν πολύ περισσότερα με τις δικαστικές υποθέσεις και αποφάσεις. Κάποιες φορές μας θεώρησαν παρεμβατικούς. Και κάποιες φορές υπήρξαν και αντιφατικές ε, παρουσιάσεις ε, στον τύπο. Όσο περισσότερο φαίνεται ότι η Γιούλεξ πάει προς ορκλήρωση της πορείας και της εντολής της, τόσο περισσότερο, τόσο περισσότερο ψύχρεμα αντιμετωπίζεται το κοσφοπέδιο και το έργο της. Για το κράτος δικαίου ξέρουμε ότι δεν είναι απλώς μια τεχνική προσπάθεια. Συνήθως απαιτεί και κοινωνικές αλλαγές. Αλλαγές στα πρότυπα και τη συμπεριφορά της κοινωνίας. Σε δέκα λοιπόν χρόνια θα ήταν ε, άδικο για τους Κωσοβάρους να περιμένουμε ότι θα έχουν αλλάξει άρδιν. Το κράτος δικαίου είναι ευρωπαϊκό μονοπάτι και δρόμος, είναι ευρωπαϊκή προσπάθεια ε, μεταμόρφωσης. Χρειάζεται πόνος, οδύνες, ε, χρειάζεται κόπος. Ε, παρόλα αυτά, μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας, ε, το αποτέλεσμα είναι καλοδεχούμενο. Αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε και στους Κωσοβάρους. Πού βρίσκεται τώρα το Κωσυφοπαίδιο. Το Κωσυφοπαίδιο βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ε, σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης, με σκαμπανεβάσματα προφανώς. Όμως, η άποψή μου είναι ότι το Κωσυφοπαίδιο έχει ενωδική πορεία. Παρόλο που υπάρχουν ε, και κάποιες οπισθοχωρήσεις, δεν είναι τα πάντα τέλεια, θα ήταν άδικο να λέμε ότι το δικοσφοπέδιο δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εμείς πιστεύουμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Και βεβαίω αυτή η μακρά πορεία προς το κράτος δικαίου είναι η ίδια ε, η πορεία προς την Ευρώπη. Και υπ' αυτήν την έννοια οι Κωσοβάροι χρειάζονται τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε υπό την μορφή της Γιούλεξ είτε άλλων ευρωπαϊκών εργαλείων. Χρειάζονται περισσότερη προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω οι νέοι, διότι ένα μεγάλο μέρος του ε, πληθυσμού του Κωσοφοπεδίου είναι 130. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του Κωσοφοπεδίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία Παπαδοπούλου για αυτή την απενημέρωση. Ήταν διεξοδικότατη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Βλέπω εδώ τον κύριο Σόλτες, ο Σόλτες, που είναι εισηγητής για το κοσυφοπαίδιο. Θέλετε το λόγο? Πολύ ωραία. Thank you, Madam for the floor. Yes, thank you. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Παπαδοπούλου για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας με πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία και απόψεις που εκφράσατε για το μέλλον της περιοχής. Έχετε παρακολουθήσει εκ του σύνταγκης, εκ του όλη αυτή τη δουλειά και εγώ την έχω παρακολουθήσει, όχι σήμερα μόνο, αλλά και από παλιά. Έχουμε παρακολουθήσει όλοι στενά την συμμετοχή σας στην εξέλιξη της ε, κοινωνίας στο Κοσφοπέδιο. Έχω κάποια ερωτήματα να σας θέσω, αν μου επιτρέπετε. μετά τη νέα εντολή, όπως αποκαλείται, που θα λάβει η χώρα τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο οι δικαστές του κοσφοπεδίου θα είναι σε θέση να αντισταθούν ε, στην πολιτική πίεση, στην παρέμβαση και στο υψηλό επίπεδο των περιπτώσεων διαφθοράς. Γιατί είναι αδιαφυσβήτητο ε, το ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ασκηθεί πιέσεις πολιτικής φύσης ή και άλλης φύσης. Σε ποιο βαθμό μπορεί η EULEX να συμβουλεύσει, να κυδεμονεύσει να, με την έννοια της προστασίας, να βοηθήσει το να ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα στο κοσφοπέδιο. Ε, Βεβαίω ήταν τεράστιο πλήγμα αυτό που συνέβη με τον Ιβάνοβιτς Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πλήρης έρευνα, αποτελεσματική, για τα περιστατικά. Πού βρισκόμαστε ως προς αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν εξελίξεις, μπορείτε να μας πείτε. Επίσης, για τη γειτονία, η EULEX θα πρέπει να δημοσιεύει εκθέσεις άπαξ τουλάχιστον για το τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η συμφωνία ε, σύμφωνα με το διάλογο Βελιγραδίου και Πρίστινας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να τηρείται ενήμερη η διεθνή κοινή γνώμη για την πρόοδο που έχει σημειωθεί ή για τα εμπόδια που παραμένουν και παρακολύουν αυτή τη διαδικασία. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το κράτος δικαίου. Το αναφέρατε. Πράγματι, είναι ένας από τους βασικότερους δείκτες, ε, βασικότερους οδηγούς για να ξαναβρει τη θέση του το στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εντολής της EULEX, διαβάσαμε κάποια άρθρα για το πρόβλημα του κράτους δικαίου εντός EULEX και εντός αντιπροσωπείας. Ποια είναι η γνώμη σας από αυτού. Και τελευταίο ερώτημα, πότε περιμένετε να αρχίσει να λειτουργεί η γέφυρα της Μητρόβιτσα στον ποταμό Ήβαρ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα ενθαρρύνει, θα αναθερμάνει τις σχέσεις μεταξύ του Κοσφοπεδίου και της Σερβίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σόλτες. Ο κύριος Κούκαν παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Ε, κυρία Παπαδοπούλου, για την πολύ αναλυτική, περιεκτική, συγκεκριμένη, αντικειμενική και δίκαιη παρουσίαση και αξιολόγηση που κάνατε για τις δραστηριότητες και δράσεις και τη δουλειά της EULEX και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το επίπεδο για εμάς που παρακολουθούμε τις δραστηριότητες από τότε που δημιουργήθηκε η Γιουλέξ εδώ και αρκετά χρόνια, ε, γνωρίζουμε ότι ε, επανειλημμένος ε, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτά που είπατε ήταν εξαιρετικά ρεαλιστικά και πολύ σωστά τα είπατε. Είναι μια μοναδική αποστολή αυτή που φέρνει σε πέραση η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κοσφοπέδιο. Τα καθήκοντα της αποστολής είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ ιδιαίτερα. Αναφέρατε ότι είναι ένα συνδυασμό τεχνικών και πολιτικών ζητημάτων και σε γενικές γραμμές οι δραστηριότητε της EU-LEX της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωση στο Κοσφοπέδιο, η οποία έχει ως στόχο να επικουρήσει ε, την ε, κοινωνία του Κωσυφοπεδίου που είναι η νεότερη χώρα στην Ευρώπη είναι μια αποστολή η ευρωπαϊκή εξαιρετικά σημαντική. Εκτιμώ τα μάλα αυτό το οποίο κάνετε και σας εύχομαι πραγματικά ε, καλή επιτυχία, τις θερμότερες ευχές μου για καλή επιτυχία και στο μέλλον. Έχω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Είπατε ότι μετά τις αλλαγές που έχουν προγραμματιστεί θα πρόκειται περί μιας απολύτως καινούρια αποστολής. Αποστολή με ποια έννοια όμως θα μειωθεί το μέγεθός της, υπό ποια έννοια θα είναι καινούρια και καινοφανή εμφανίσει η αυτή. Δεύτερο ερώτημα. Η EULEX είχε πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση και τους υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους. Αυτό δεν ισχύει πάντοτε στον, στο παρελθόν. Ενίοτε ασκούσαν πολύ κριτική και δεν χρησιμοποιώ καθόλου διπλωματική γλώσσα, αλλά ενίοτε έλεγαν ότι η EU διατάζει και περιμένει από εμά να τα εφαρμόζουμε. Ε, ποια είναι η κατάσταση τώρα. Επίσης χρησιμοποιήσατε τον ενδιαφέροντα όρο διαχείριση των προσδοκιών, management of expectations. Πράγματι, η EU-Lex απολαμβάνει του σεβασμού ε, που τρέφει στο πρόσωπό της ο πληθυσμός στο κοσφοπέδιο, όμως σε πολλές από τις επισκέψεις μου στο κοσφοπέδιο ακούσαμε πολύ βιαίως επικριτικές παρατηρήσεις από μη κυβερνητικούς οργανισμούς σε βάρος που καταφέρονταν εναντίον ε, της EULEX. Ανέκαθεν εμείς υπερασπιζόμαστε το ρόλο και τις δραστηριότητές της. Μερικές φορές όμως ήταν εξαιρετικά λυπηρό να ακούμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις γιατί δεν εξέφρασαν μια αντικειμενική και δίκαιη άποψη για την EULEX. Έχετε λοιπόν εμπειρία από τη συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις γιατί ο ρόλος και η δράση αυτών και αυτά που λένε οι ΜΚΟ είναι πράγματα εξαιρετικά σημαντικά. Είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει, που έχει ειδικό βάρος στην κοινωνία του κοσφοπεδίου. Ήθελα να κάνω και μια άλλη ερώτηση που την έθεσε ο κύριος Σόλτες και εγώ θα ήθελα να μάθω για τη διερεύνηση του της δολοφονίας του Ιβάνοβιτς γιατί ήταν μια πολύ δραματική στιγμή κατά την οποία διαταράχθηκε ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Τέτοιου είδους περιστατικά, τέτοιου είδους συμβάντα μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά ενδεχομένως μόνο εφόσον υπάρξει πλήρης διερεύνηση και χυθεί άπλετο φως. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν τώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Σόλτες έθεσε όλα τα επίκυρα ερωτήματα, τα πολύ σκόπιμα και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις απαντήσεις που θα δώσετε. Και συμπερασματικά θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή σας σε δύο σημεία. Πρώτον, εκτιμώ ιδιαίτερο στο έργο της EULEX. Είναι απαραίτητο για όλους εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Πρέπει όλοι να τη βοηθήσουμε την EULEX και να τη στηρίξουμε, να καλύψουμε τις ανάγκες σας, γιατί κάνετε καταπληκτικά πράγματα για την κοινωνία στο κοσφοπέδιο. Αυτό καταρχάς. Μιλήσατε για το μέλλον. Όμως, Ο τρόπος με τον οποίο μιλήσατε για το παρελθόν είναι πάρα πολύ εύγλωτος για τις νέες πτυχές και προοπτικές της μεταρρυθμισμένης αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσφοπέδιο. Ευχαριστούμε ο κύριος Μαυρίδης παρακαλώ. Um, Κυρία Παπαδοπούλου, θα μιλήσω ε, ελληνικά, τη μητρική μου γλώσσα. Αν χρειάζεστε διερμηνία μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά. Θα ξεκινήσω και εγώ λέγοντας ότι θέλω να σας συγχαρώ. Θέλω να σας συγχαρώ για την εργασία που κάνετε στο Κόσοβο ε, και όντως συμμερίζομαι για αυτά που έχετε πει ότι πρόκειται για μια ίσως από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις από στα Δυτικά Βαλκάνια. Το πρώτο μου ερώτημα όμως είναι εκεί που πιστεύω ότι κάνατε και μια σημαντική δουλειά. Είναι σε αυτό που ονομάζουμε war crimes. Μπορείτε να μας πείτε τι θα είναι η επόμενη μέρα, για παράδειγμα, θα υπάρχει ε, δραστηριότητα του International Criminal Court ή θα αφήσουμε το Κόσοβο μόνο του. Whatever that means. Ε, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και για άλλες περιπτώσεις και θα δείτε στη συνέχεια τι εννοώ για εγκλήματα πολέμου. Το δεύτερο είναι ότι, ε, όπως σωστά έχει λεχθεί, τα αποτελέσματα δεν πρέπει να κρίνονται μόνο με το σενάριο που βλέπουμε στο έδαφος, αλλά πώς θα ήταν η κατάσταση αν δεν υπήρχε το Ulex, όντως. Ωστόσο, ένα συμβάν που δεν τέθηκε σήμερα και νομίζω έχει αμαυρώσει ε, την, την, το όλο rule of law in Kosovo είναι η απαγωγή των έξι καθηγητών, δασκάλων, οι οποίοι ήταν τουρκικής εθνικότητας, απήχθηκαν και κανένας μας δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα ποια ήταν η μοίρα τους. Δεν θα αρχίσω να μπω στη διαδικασία ότι ο ίδιος Ομπτουσμάν του Κόσοβο μίλησε για κατάφορη παραβίαση του rule of law. Αλλά τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι και μάλιστα θα σας πω επειδή έχουν περάσει και αρκετοί μήνες είναι ασφαλές να σας πω ότι σας δόθηκε πληροφορία ότι αυτά τα έξι πρόσωπα κρατούνταν παράνομα στο παλιό αεροδρόμιο και όχι στο νέο αεροδρόμιο όπου ψάξατε. Θα ήθελα να μας δώσετε μια πληροφορία γύρω από αυτό. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η τύχη τους. Ε, και τελειώνω με μόνο μία παρατήρηση. Όταν σας παρακολουθούσα και μου άρεσε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήραμε πρωτοβουλία για το rule of law, ειδικά σε σχέση με την απόδοση της δικαιοσύνης, διερωτώ με αν όλοι μας, και αυτό δεν είναι για σας, είναι να τα ακούσουμε όλοι μας εδώ, κατά πόσον θα πρέπει κάτι παρόμοιο και ανάλογο να προσαρμόσουμε και στην περίπτωση της Τουρκίας του Ερτογάν, εκτός αν πιστεύουμε ότι εκεί υπάρχει απονομή της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ που με ακούσετε. Thank you, Mr. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Μαυρίδη. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Εάν όχι, να δώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ε, σημαίνει πολλά για όλους εμάς την Γιούλεξ. Να ξεκινήσω από τα βασικότερα, την υπόθεση Βάνοβιτς που έχει να κάνει τα γεγονότα. Ε, ενημερώθηκε η μονάδα μας ε, αμέσως από την αστυνομία του Κοσφοπεδίου παρακολουθούμε την υπόθεση κοιτάζοντας τι ακριβώς κάνει η αστυνομία στο Κωσφοπέδιο και κοιτάζουμε επίσης να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της επίσημης αστυνομίας του κοσυφοπέδιο και των σερφικών αρχών στο προσωπικό μας την Ulex φροντίσαμε ήδη να υπονηθεί αποτίμηση των δραστηριοτήτων της αστυνομίας του Κοσμοπεδίου. Τη μοιραστήκαμε μάλιστα μαζί τους, πήραμε τα σχόλιά τους για το τι ενέργειες ακολούθησαν για την έρευνα αυτή και θα κοιτάξουμε να χρησιμοποιεί η έκθεση αυτή για τους σωστούς σκοπούς. Την έρευνα πάντως ανέλαβε η κεντρική υπηρεσία στην Πρίστινα, διότι στο βορρά δεν υπήρχε αρκετή τεχνογνωσία για να αντιμετωπιστεί μια τόσο περίπλοκη υπόθεση. Τώρα έχει αναλάβει η Πρίστινα οι αστυνομικοί τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων στην Πρίστινα συνεργάζονται με του ε, συναδέλφου του στο Βορρά, αλλά η συνεργασία κάποιε φορέ έχει δυσκολιούλε. Δεν υπάρχει καμιά φοβερή μεγάλη εξέλιξη που να είναι ορόσημο, αλλά την ευθύνη την έχει η Κωσοβάρικη αστυνομία και εμείς ως Γιούλεξ έχουμε συναντήσεις με προσώπους ε, της Σερβικής Αστυνομίας και της αστυνομίας ε, του Κοσφοπεδίου. Αυτά περί της συγκεκριμένη υπόθεσης. Τώρα για τις διάφορες ε, παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Σόλτες για την Ιούλεξ. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι η Ιούλεξ εφαρμόζει με θρησκευτική ευλάβεια πολύ αυστηρός όλους τους κανόνες που ισχύουν για να αντιμετωπιστούν, να καλυφθούν τέτοιε ε, υποθέσεις. Είναι σαν το Ευαγγέλιό μας αυτό, στο οποίο έχουμε ορκιστεί. Και ως αποστολές πρέπει να πω ότι έχουμε μηδενική ανοχή προς τη διαφθορά ή την πολιτική, τον πολιτικό παρεμβατισμό. Οι έρευνε που γίνονται στι Βρυξέλλε, όσο έχει στη Γιούλεξ, στι Βρυξέλλε, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι αρκετέ. Είμαι πεπισμένη ότι όλα τα ζητήματα ε, εξετάζονται επαρκώς και ο κώδικας συμπεριφοράς υποχρεώνει τα μέλη μιας αποστολής να συμπεριφέρονται με τα πρότυπα συμπεριφοράς ε, που είναι τα δέοντα, ιδίως μια αποστολή όπως αυτή στο Κωσφοπαίδιο. Πάντως, ε, δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε και το εξής, το τεκμήριο αθωότητας. Ε, υπήρξαν κάποιες κατηγορίες εδώ που ε, έδειξαν ότι εν τέλει ήταν ε, βάσιμε. βασίζοντας σε πραγματικά γεγονότα. Αυτό έπληξε το ηθικό τη αποστολή και αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Η αποστολή πρέπει να γίνεται σεβαστή. Και είμαι απολύτως πεπισμένη ότι οι συνάδελφοί μου διέπονται από πλήρη ακαιρεότητα. Αν κάποιο έχει κάνει κάτι το επιλήψιμο, ο κώδικας συμπεριφορά ή οι κανόνες της αποστολή θα ισχύσουν, θα εφαρμοστούν. Όμως Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου και υπεύθυνοι είναι και έντιμοι. Άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν. Με τρόπο επαγγελματικό και σε συνθήκες αρκετά δύσκολες. Οι σχέσεις με τους ντόπιου. Όπως είπα προηγουμένως και αρκετά γενικόλογα, οι διαθέσεις προς τη Γιούλεξ περνάνε από διαφορετικές φάσεις. Έχω μιλήσει με πολλούς από μη κυβερνητικέ οργανώσει στο κοσφοπέδιο και πολλέ φορέ είναι ιδιαίτερα επικριτικοί, διότι περίμεναν να του δώσουμε τον ουρανό μετάστρα και δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Δεν μπορούσαμε, κανεί δεν μπορούσε. Και σε άλλα μέρη, όχι μόνο στο κοσφοπέδιο, και σε άλλα μέρη στον κόσμο, πολλέ φορέ οι ντόπιοι κοιτάνε τη διεθνή δύναμη περιμένοντα να του λύσουν τα προβλήματά του. προβλήματα που πρέπει να λύσουν οι ίδιοι. Ένα πράγμα που προσπαθώ να καταστήσω σαφέ στο Κοσφοπέδιο, εδώ και δύο χρόνια που βρίσκομαι εκεί, είναι ότι η Ulex δεν πήγε εκεί για να υποκαταστήσει την οικοδόμηση θεσμών στο Κοσφοπέδιο, να του βοηθήσουμε, να του συνδράμουμε, να του οδηγήσουμε, να είμαστε στη διάθεσή του. Όμω μετά τι δικέ του επιλογέ που να κάνουν, τη δική του θέση να διεκδικήσουν, τη δική του ζωή και το δικό του μέλλον. Κάποιες φορές ε, βρίσκονται σε σύγχυση. Τώρα που η Ulex σιγά σιγά αποχωρεί, όλοι κάπω έχουν αγχωθεί για το κενό που θα αφήσει πίσω Εγώ τους καθησυχάζω ότι βρίσκεται η Πατιαρμοστία, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γιούλεξ με διαφορετική μορφή. Αλλά πρέπει να αποδεχθούν ότι είναι δική τους ευθύνη. Εκείνη είναι η υπόλογη προς το δικό τους λαό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ε, έχουμε ακόμη σκαμπανεβάσματα, διότι κάποιες φορές η Γιούλεξ ε, δίνει την εντύπωση δεν τους συμπαθεί πολιτικά. Γιατί, όπως έλεγα, οι δράσεις μας έχουν πολιτικές συνέπειες στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτό σε κάποιους δεν αρέσει. Όμως τα πράγματα έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ, προφανώς. Και πρέπει να πω ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με όλους. και με τις αρχές τους και με τις κυβερνητικέ τους οργανώσεις και κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, των ικανοτήτων μας και της εντολής μας, ό,τι αφορά τη νέα αποστολή. Δεν θα περιοριστεί μόνο σε αριθμούς πολλές από τις βασικές μας δραστηριότητες επιστρέφουν ε, στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα συμμετέχουμε στον σχεδιασμό νομοθεσία ή στο Δικαστικό Συμβούλιο του Κωσφοπεδίου. Αυτά θα τα αναλάβουν ε, οι υπεύθυνοι του ΙΕ. Θα έχουμε ακόμη πολλές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπως οι διορθώσεις, η παρακολούθηση υποθέσεων και φακέλων που είχαμε αρχίσει ήδη να κοιτάζουμε με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και όλα αυτά θα γίνουν σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο και το ΝΟΕ. Αλλά έχουμε ακόμη την τεχνογνωσία, θα την παράσχουμε απλώς σε στενή συνεργασία με την με την EUSR. Ε, Ίσως όχι τόσο γρήγορα όσο περιμέναμε, πάντως τα πράγματα προχωρούν. Τώρα για το πώς χειρίζονται οι δικαστές τις υποθέσεις. Όπως σε κάθε σύστημα υπάρχουν καλοί, κακοί δικαστές, μέτρη, λογικό είναι αυτό. Αλλά η παρουσία της Γιούλεξ είναι αποτρεπτικός παράγοντας και μόνο το γεγονός ότι παρακολουθεί, ότι παρατηρεί, ότι καταγράφει τα πράγματα σε ε, φέρνει αποτέλεσμα. Είμαι πεπισμένη, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον βεβαίω, δεν είμαι μάντης, ούτε μπορώ να σας πω ότι όλα θα γίνουν τέλεια, αλλά είμαι πεπισμένη ότι αυτός ο δρόμος θα συνεχίσει να ακολουθείται. Είμαι πολύ πεπισμένη γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα πολέμου, το δικαστήριο της Χάγης είναι ανεξάρτητος θεσμός και εργάζεται ανεξαρτήτως οποιοδήποτε. Δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι θα κάνουν τη δουλειά του στο μέλλον όπω την κάνουν τώρα. Πολλέ ε, υποθέσει πολέμου ε, ε, έχουν εξεταστεί από τη Γιούλεξ. Έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώ. Πολλέ έχουν ήδη αποσταλεί έτοιμε με την ανάκριση ολοκληρωμένη στου υπεύθυνου και θα τι παρακολουθεί η Γιούλεξ και στο μέλλον στην εκδίκασή του και νομίζω η προσπάθεια αυτή να τιμωρηθούν ω το δυνατόν περισσότερα εγκλήματα θα συνεχιστεί. Σε ό,τι αφορά το κοσφοπέδιο ε, και την ε, συζήτηση στο Κοινοβούλιο, αυτό συζητήθηκε μόλις προχθές και προκάλεσε πολιτική καταιγίδα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συζήτησης στο Κοινοβούλιο, γιατί έγινε μόλις προχθές, αλλά θα ε, φτιάξουν επιτροπή για να διερευνήσει το τι συνέβη. Έχουν αναλάβει λοιπόν την απαραίτητη πρωτοβουλία. Πρόεδρος, ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε για όσα κάνετε για την Γιούλεξ και σας ευχόμαστε καλή τύχη. Ολοκληρώνεται η ανταλλαγή μα και η συζήτησή μα σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ και εσά. Ευχαριστούμε για την απενημέρωση. Θα μείνουμε σε επαφή. Σε οποιαδήποτε θέση. Δύο λεπτά διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με, το σημείο 18. Ενημέρωση σχετικά με την ε, ε, αποστολή παρατήρησης εκλογών στο Λίβανο. Η αποστολή έλαβε χώρα από τις 3 έως τις 8 Μαΐου. Κυριακή 6 Μαΐου έγιναν οι εκλογές, 10 χρόνια μετά τις προηγούμενες εκλογές, το 2009 μάθαμε ότι η χώρα έχει θεσπίσει νέο εκλογικό νόμο πριν από ένα χρόνο και πολλές από τις συστάσεις που είχε κάνει η προηγούμενη αποστολή των παρατηρητών είχαν ληφθεί, έχουν ληφθεί υπόψη. Δυστυχώς η προσέλευση είναι χαμηλότερη από την προσέλευση το 2009 να καλωσορίσω την κυρία Ελένα Βαλενθιάνο, που ήταν επικεφαλής της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών στον Λίβανο. Να καλωσορίσω τον κύριο Χωσέ Ιγνάθιο Σαλαφράγκα, πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Βαλενθιάνο, να μας μιλήσετε για την Αποστολή καταρχάς και μετά να πάρει το λόγο ο κύριος Σαλαφράγκα που θα μας πει και αυτός δύο λόγια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, η εκλογική αποστολή παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκλογές στο Λίβανο διοργανώθηκε, έλαβε χώρα. Από τα τέλη Μαρτίου είμαστε παρόντες, δηλαδή από τα τέλη Μαρτίου δουλεύουμε για αυτή την αποστολή παρατήρησης της εκλογικής διαδικασίας με πολύ σημαντική ομάδα ανθρώπων που στείλαμε σε όλη τη χώρα αλλά και στην πρωτεύουσα με τους συνήθεις εμπειρογνώμονες για, ως παρατηρητές για την εκλογική διαδικασία. Πρόκειται για εξαιρετική δουλειά κατά την άποψή μου από τεχνική σκοπιάς, ε, μια δουλειά που επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώσει ε, τη σημαντική της παρουσία η οποία ξεχώρισε και την οποία εκτίμησαν δεόντως όλοι οι συνομιλητές μας. Όπως είπε και η αξιότιμη κυρία Πρόεδρος, ήταν μια ευκαιρία αυτή να γίνουν εκλογές με έναν καινούριο εκλογικό νόμο ένα νόμο τον οποίο εμείς είχαμε αξιολογήσει, είχαμε εμείς συστήσει και τον είχαμε συμβουλεύσει να υιοθετηθεί και να ενσωματηθεί μαζί με άλλους πολιτικούς παράγοντες ένα εκλογικό νόμο που ενσωμάτωνε πολύ σημαντικά στοιχεία πολιτικής αλλαγής. Και καταρχάς συμπιωνόταν πρόοδος γιατί πάμε προς ένα πιο αναλογικό σύστημα. Ενσωματώνεται η ψήφος των Λιβανέζων που ζουν στο εξωτερικό και διαφυλάσσεται περισσότερο το απόρριτο της ψήφου από τη στιγμή που ήταν προηγουμένως εκτυπωμένα ψηφοδέλτια για τους ψηφοφόρους. Αυτές ήταν οι βασικές μας συστάσεις και τροποποιείται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τροποποιήθηκε όχι μόνο η εκλογική νομοθεσία, αλλά και ο τρόπος του ψηφίζει, να θέλετε, η, η εκλογική κουλτούρα και συνήθεια των Λιβανέζων. Η ημέρα λοιπόν ε, των εκλογών, της ψηφοφορίας, ε, κύλησε πολύ ήρεμα, πολύ ειρηνικά, εκτός από πολύ λίγα συμβάντα. Όλοι οι παρατηρητές μας ανέφεραν ότι πρόκειται για μια διεξαγωγή μιας ομαλούς εκλογικής διαδικασίας, παρά ε, τις λίγες κριτικές που προέκυψαν τις επόμενες μέρες, οι οποίες κόπασαν σιγά σιγά. Επομένως, η αξιολόγησή μας είναι ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε ήρεμο κλίμα και γι' αυτό κάθε φορά που γίνεται αυτό ενισχύεται η αξιοπιστία τους. Πολύ αποτελεσματικά ήταν τα ψηφοδέλτια, εκλογικοί κατάλογοι, δεν έγιναν παρατηρίες, παρατυπίες αξιοσημείωτες. Ορισμένοι υποψήφοι που δεν κατάφεραν να κερδίσουν μία έδρα παραπονέθηκαν ότι οι διαδικασίες δεν ήταν αξιόπιστες, όμως και αυτά τα σχόλια τελικά καταλάγιασαν. Ορισμένα στοιχεία της προεκλογικής εκστρατείας και του πολιτικού συστήματος στο Λίβανο μας ανησυχούν βεβαίως και τους συνομιλητές μας αλλά και τους υποψηφίους και τα πολιτικά κόμματα που παρίστανται και ε, βάζουν υποψηφιότητα για τις εκλογές. Έχουμε να κάνουμε με τον έλεγχο της χρηματοδότησης, τα τεράστια ποσά χρηματικά που κινούνται γύρω από τις εκλογές. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες ήταν τεράστια τα ποσά που διακινήθηκαν για την προεκλογική εκστρατεία η δυνατότητα της Επιτροπής Εκλογικής Παρατήρησης, η οποία ήδη υπάρχει και δραστηριοποιείται, να ελέγξει όλο αυτό τον όγκο χρηματικό ποσόν που κινούνται, είναι απολύτως μηδενική. Είναι μια Επιτροπή Παρατήρησης της εκλογικής διαδικασίας, η οποία εξαρτάται άμεσα από την κυβέρνηση και έχει πολύ μικρή δυνατότητα να διερευνήσει τις πηγές χρηματοδότησης των διαφόρων υποψηφίων. Μία από τις συστάσεις μας στην έκθεση άλλωστε την προκαταρκτική που συντάσσουμε είναι να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες ερευνητικές και ελέγχου εκλογικού σε αυτή την Επιτροπή. Να έχει δικό της προϋπολογισμό, να έχει αυτονομία και ικανότητα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη μας, που δεν ε, τηρήθηκε, είναι να ενσωματωθούν οι γυναίκες στην πολιτική εξουσία, να έχουν την δυνατότητα να εκλεγούν ήταν και μία από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2009. Παρόλο δηλαδή που είχαμε πολύ περισσότερες υποψήφιες από το 2009, μόνο έξι γυναίκες εξελέγησαν στο Λιβανέζικο Κοινοβούλιο. Είναι από τα κοινοβούλια που έχουν τη μικρότερη εκπροσώπηση γυναικών στον κόσμο σε μία χώρα στην οποία οι γυναίκες είναι εξαιρετικά δραστήριες και καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας και της, εκλογικής, ε, ε, της ημέρας των εκλογών είδαμε ότι οι γυναίκες είναι πρωταγωνίστριες και στις προ εκλογική εκστρατεία και στη διαχείριση τη εκλογική διαδικασία. Όμω είναι πολύ δύσκολο να εκλεγούν στι θέσει, στα αξιώματα και αυτό είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει και το θέτουμε συνεχώ στου συνομιλητέ μα, στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, στου πολιτικού φορεί κτλ. Τώρα, η ενσωμάτωση τη ψήφου των ομογενών των ε, Λιβανέζων του εξωτερικού ήταν εξαιρετικά σημαντική και σε επίπεδο συμβολικό και αλλού. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την παρατήρηση των εκλογών στις διάφορες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου μπόρεσαν οι Λιβανέζοι να μεταβούν και να ψηφίσουν. Είχαμε απόλυτα έλεγχο για το πώς ανοίγουν οι κάλπες στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού για να ψηφίσουν οι Λιβανέζοι του εξωτερικού και άρα έχουμε μια πλήρως κατοχυρωμένη, διαφανή, ειλικρινή και σωστή διαδικασία σε αυτό το επίπεδο. Τώρα το άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο της Επιτροπής είναι η πρόσβαση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι ή δεν έχουν αρκετά χρήματα ή είναι ξένοι προς το σύστημα των ε, λιβανέζικων πολιτικών κομμάτων. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στο Λίβανο, τα τηλεοπτικά κανάλια, το κάθε ένα σχετίζεται άμεσα με κάθε ένα από τα κόμματα τα μεγάλα που παρουσιάζονται και βάζουν υποψηφιότητα και που κατεβαίνουν στις εκλογές. Άρα πάρα πολλά από τα μέσα επικοινωνίας ακολουθούν την εξτροτεία των μεγάλων κομμάτων. Άρα ισότητα των ευκαιριών στην, ε, ε, στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια παρουσία είναι κάτι το οποίο δεν κατοχυρώνεται σε καμία περίπτωση. Συμπερασματικά λοιπόν, γιατί αυτά είναι και τα τελευταία στοιχεία που μπορώ να κομίσω ε, από τότε που ήρθα από τη Βηρητό. Συμπερασματικά, ανάγνωση των αποτελεσματών όπως είπε και η Πρόεδρος, πράγματι η προσέλευση ήταν εξαιρετικά χαμηλή, χαμηλότερη από ότι το 2005 και το 2009, όχι θεαματικά πιο χαμηλή, 44% ε, το 2005, αλλά ήταν πιο χαμηλή από ότι το 9. 49,2% η προσέλευση φέτος. Σε μια χώρα όπου δεν είχαν γίνει εκλογές για 10 χρόνια, φαίνεται αντιφατικό τώρα που τους δόθηκε ευκαιρία τόσοι λίγοι να εμφανιστούν να ψηφίσουν. Το σίγουρο είναι ότι η δημοκρατία είναι μια άσκηση η οποία βελτιώνεται κάθε μέρα. Δηλαδή όσο περισσότερο ασκεί κανείς δημοκρατία, τόσο περισσότερο ασκείται σε αυτήν και την κάνει όλο και καλύτερα. Τώρα ως προς τα αποτελέσματα, εν συντομία να πω δύο λόγια και φαντάζομαι ότι ο συνάδελφος, ο πρόεδρος της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Σαλαφράγκα, θα πει περισσότερα. Άλλωστε είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον κύριο Σαλαφράγκα και θέλω να το ευχαριστήσω θερμά και εκείνον και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω να συμφωνεί μαζί μου το χαρίρι ε, δέχθηκε πλήγμα περιορισμένο, συνεχίζει να εκπροσωπεί την πλειοψηφία, να αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα Σουνιτών στο Λιβανέζικο Κοινοβούλιο έχει μια συμβολική αξία σημαντική. Ο Μασνούκο, ο Υπουργό Δικαιοσύνη, μα έλεγε ότι στι μικρέ χώρε τα σύμβολα είναι σημαντικά. Και όντω το ε, είναι σημαντικό πολιτικό σύμβουλο και ε, διατηρεί τη δύναμή του. Οι Λιβανέζικε δυνάμει κατοχυρώνουν τη δύναμή του και η αναλογικότητα ευνόησε αυτό το κόμμα, Λιβανέζικε δυνάμει και η Ουμλαντ διατηρεί τα ποσοστά της και άρα την επιτορή της. Η Χεσμολά και η Αμάλ ανέβηκαν αλλά όχι τόσο πολύ όσο λέει ο τύπος της δύση, όπου τα πρωτοσέλιδα έλεγαν ότι είχε πολλά θριάμβευσε στις εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι ανέβηκαν τα ποσοστά της, αλλά όχι τόσο. Υπάρχει μεγάλη συνένεση στο γεγονό ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας. Και το σύνολο του πολιτικού φάσματος στο Λίβανο μας το είπε αυτό, να μην γίνει τίποτα που θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας. Θα υπάρξει κυβέρνηση ενότητα. Πάρα πολλές συμβαστικές λύσεις πρέπει να ε, επιτευχθούν για να γίνει κάτι τέτοιο. Επομένως θα έχουμε προεδρία του ΑΟΥΝ με το Χαρίρι στην κυβέρνηση. Πολύ σημαντικό ρόλο θα διαδραματίζει το στρατόπεδο των χριστιανών. Τώρα, Ούτε η κυβέρνηση του Ισραήλ, ούτε η κυβέρνηση των ΙΠΑ δεν μπορούν να υποδίσουν μια χώρα αφόσον θέλει να πορευθεί αυτόνομα με όλες τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται. Ε, υπάρχει επιθυμία στη χώρα αυτή να ξεφύγουν από τη μόνιμη επιτροπή των μεγάλων χωρών, των γειτονικών χωρών. Ένα μικρό συμβάν έγινε με μέρος της, των ψήφων της Οργανωμένης Κοινοτίας των Πολιτών όταν έκλεισαν οι κάλπες. Μία υποψήφια θεωρούσε ότι έχει την έδρα, αλλά μετά με την εκ νέου καταμέτρηση φάνηκε ότι δεν την κερδίζει την έδρα με διαφορά χιλίων ε, ψήφων περίπου. Μία πολύ γνωστή εκπρόσωπος της Οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών, δημοσιογράφος, συγγραφέας και που αρθρογραφεί και το καθεξής. Τελικά δεν κέρδισε την έδρα και συναντήσαμε και ρυθμίσαμε τα πράγματα. Η χριστιανική ψήφος είναι η ψήφος της ανώτερης, αν θέλετε, τάξης, της πιο εκπαιδευμένης, της πιο μορφωμένης και αυτή είναι και η ψήφος προς τους εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Γενικά έχουμε θετική αντίληψη για την εκλογική διαδικασία. Θα παραμείνουμε στη Βηρητό μέχρι τις 7 Ιουνίου, περίοδο ε, κατά την οποία λήγουν οι ενστάσεις και στη συνέχεια θα καταρτήσουμε την τελική μας έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαφράγκα για τη συνεργασία και τη δουλειά του και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την πρέσβειρά μας στην Βηρητό, την Κριστίνα Λάρσεν, για την εξαιρετική τη συνεργασία και στον Τζανφριάν Κομποκίγιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που μας συνόδευσε, που μας πλαισίωσε, που μας έδωσε όλα τα μέσα και τις δυνατότητες, μας βοήθησε και μας επέτρεψε να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα που προέκυψαν επί τόπου. Μια εξαιρετική αποστολή σε μια πραγματικά εξαιρετική χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Βαλενσιάνο. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω στην ανάλυση που μας παρουσίασε η Έλενα Βαλενθιάνο και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα πολύ απλά να πω ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε την ευκαιρία να κάνει μια αποστολή και να επισκεφθεί τη Διεθνή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών που είναι ανεπτυγμένη στο νότιο Λίβανο για να μπορέσει να σπιγμωματρήσει την γαλάζια γραμμή και να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Ήταν θετική η εμπειρία μας ότι παρά τις εντάσεις που βιώνουν στην περιοχή και παρά τις μεταναστευτικές πιέσεις τις πολύ σημαντικές από τις οποίες υποφέρει η χώρα με 1,5 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες στα εδάφη της, η εκλογική διαδικασία διεξήχθηκαν με, σε ομαλές συνθήκες, με ομαλό τρόπο και ήρεμο τρόπο, όπως υπογράμμισε και η κυρία Έλενα Μπαλανθιάνο. Ο Λίβανος και η σταθερότητά του είναι ένα στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό στην Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει παρακολουθεί στην εκλογική διαδικασία και το 2005 και το 2009. Πράγματι, η προσέλευση, η συμμετοχή στις εκλογές ε, δεν ήταν τόσο υψηλή όσο το 2009, ωστόσο αν τη συγκρίνουμε με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα ή στις δημοτικές εκλογές ε, που έχουμε εμείς στην Ευρώπη ποσοστά του στυλ 33% ε, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι και στο Λίβανο ήταν καταστροφή η συμμετοχή στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, εμεί ω μέλη του, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκοληθήκαμε στην αποστολή παρατηρητών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαστήκαμε άψογα με την κυρία Βαλενθιάνο και λόγω των συνθήκων της χώρας αυτής και λόγω ε, του νέου εκλογικού νόμου δεν είχαν γίνει εκλογές στη χώρα αυτή για 9 χρόνια. Δεν νομίζω ότι κανεί θα ήθελε από εμάς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνουμε στις θέσεις μας για μια ολόκληρα χρόνια χωρίς να ξαναμιλήσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί ε, και να αποφαθούν για τη δουλειά μας. Ένα σημαντικό στοιχείο που υπογράμμισε και η αποστολή των παρατηρητών είναι το εξή. Επειδή πέρασε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και επειδή πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα, πάνω από 700.000 νέοι ψηφοφόροι ψήφισαν για πρώτη φορά και αυτό το ποσοστό μεγάλωσε. Ε, δηλαδή αυτό μεγάλωσε το ποσοστό των ψηφοφόρων που απήχαν από τις εκλογές. Γιατί 700.000 ούτως ή άλλως ήρθαν ε, για πρώτη φορά από αυτούς. Άρα περισσότεροι από τους προηγούμενους δεν ε, ψήφισαν. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών η χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατιών, η στήριξη και η βελτίωση των δυνατοτήτων και μέσων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Εποπτείας της εκλογικής διαδικασίας. Είναι θέματα που θέσαμε. Είναι σημεία στα οποία φυστήσαμε την προσοχή. Υπογραμμίσαμε την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλει προς την κατεύθυνση που ανέφερε η Έλενα, προς την σταθερότητα, τη σχετική σταθερότητα στη χώρα. Γιατί η σταθερότητα στο Λίβανο είναι μια σταθερότητα όχι επισφαλή, σάλα αποτελεί απεικόνιση του πολύχρωμου μοσαϊκού ε, με τις πολλές και διαφορετικές ψηφίδες που συγκροτούν τη λιβανέζικη κοινωνία. Ε, ε, κοινωνία. Πήγαμε προς ένα πιο αναλογικό σύστημα. Είχαμε ψηφοδέλτια τυπωμένα με τα ονόματα των υποψηφίων, πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές προόδοι και επιτέματα σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Τώρα, η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι οι εκλογές ήταν καλά οργανωμένες, διεξήχθησαν σε συνθήκε ομβαλότητας, ε, οι πολίτες επέδειξαν πρακτικό πνεύμα, ρεαλιστικό υπήρχαν αμφιβολίες για την κατανόηση από πλευράς της λιβανέζικης κοινή γνώμης του εκλογικού νόμου, ο οποίος ήταν κάπως περίπλοκος. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι δεν έχουν σημειωθεί τρομακτικές και κολοσιές αλλαγές, αλλά καλύτερα είναι τα πράγματα και μπορούν να διατηρηθούν σταθερά σε μια χώρα τόσο δύσκολη, σε ένα περιφερειακό πλαίσιο τόσο περίπλοκο και άρα φεύγουμε από τη χώρα κρατώντας θετική εντύπωση και εκφράζουμε την επιθυμία να διεγείρουμε το ενδιαφέρον των νέων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν περισσότερο στο δημόσιο γίγνεσθε Ορισμένοι συνομιλητές μας παραδέχθηκαν ότι στους εκλογικούς τους καταλόγους δεν είχα συμπεριλάβει ούτε μία γυναίκα και μάλιστα ε, είχαν έρθει σε δύσκολη θέση όταν έπρεπε να το παραδεχθούν αυτό γιατί ήταν εκπρόσωποι και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό των Υπουργών Εσωτερικών που εποπτεύει την εκλογική διαδικασία, με τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας Εκλογών, ε, όλες αυτές οι συναντήσεις μας άφησαν με θετικές εντυπώσεις και νομίζουμε ότι και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς κάναμε την καλύτερη δυνατή εντύπωση. Ε, τονίσαμε τη σημασία, τη σημασία της συμφωνίας σύνδεσης, τα προγράμματα που έχουμε, που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την οικονομική πρόοδο, τη χρηστή διακυβέρνηση. Η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, έχει υψηλό δημόσιο χρέος 140%, έχει ανεργία ε, μεγάλη και αυτό οξύνεται με την παρουσία προσφύγων από τη Συρία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει γενικότερη βούληση να υπερπηδηθούν οι δυσκολίε και να συνεχίσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Τέλο, υπογραμμίζουμε το γεγονό ότι χρειάζεται να ενισχυθούν οι σχέσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μεταξύ δύο κοινοβουλίων και να αναπτύξουμε την τεχνική συνεργασία με το Κοινοβούλιο του Λιβάνου. Να ευχαριστήσω την κυρία Βαλενθιάνο για την υποδοχή και τη φιλοξενία, για τη στήριξη που μας προσέφερε. Ε, σε εμά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι οι βουλευτές είδαν πόσο ε, καλά συνεργαζόμαστε και αυτό είναι αναπόδραστο και είναι ευκταίο και επιθυμητό να συνεργαζόμαστε ομαλά και άψογα μεταξύ ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωση για την παρατήρηση της εκλογική διαδικασίας. Να ευχαριστήσω θερμά τις γραμματείες που ε, ακούραστες ήταν και έφεραν σε πέρα και ρύθμισαν όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και ελπίζω η αποστολή αυτή να έχει το θετικό αντίκτυπο που περιμένουμε. Να συγχαρώ όλους και να ευχαριστήσω όλους για τη δουλειά τους και να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία η οποία στήριξε με υποδειγματικό τρόπο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στην αποστολή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Εγνάσιο. κυρία Ματίας θέλει το λόγο. Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με, την... με τις χώρες μας ΡΕΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Βαλενσιάνο Ξαλαφράκα για τη δουλειά τους. Συμμερίζομαι και συμφωνώ με το περιεχόμενο των όσων είπαν. Να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας από τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου και να επισημάνω ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσυπογράφω πλήρωση όσα είπε η Έλενα Βαλενσιάνο και την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου όπου προέδρευε ο κ. Σαλαφράγκα. Απλώ να προσθέσω ένα σημείο που έχει να κάνει με τη μορφή με την οποία οι δύο αντιπροσωπείες, η μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άλλη του Ευρωκοινοβουλίου, εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους σε ένα πλαίσιο αρκετά λεπτό ε, πολιτικών δυσκολιών εδώ και μια χρόνια. εγκρίθηκε όχι απλώς ένας νέος εκλογικός νόμος, δύο προπολογισμοί και ο πολιτικός βίος πήρε μπρο σε ένα τοπίο αρκετά δύσκολο για το λιβανέζικο λαό. Για τα τελευταία χρόνια έχουν υποδεχτεί, όπως ξέρουμε, τόσους ε, πρόσφυγες από τη Συρία. Σε συνθήκες που δεν είναι και πιο απλές, δεν έχουν τόσες πολλές δυνατότητες και έχουν φανεί ιδιαίτερα γενναιόδοροι. Γι' αυτό λοιπόν οι δύο αυτές ποστολές εκπλήρωσαν το ρόλο τους με τρόπο εξαιρετικό θεωρώ και οι δύο επικεφαλής αντιπροσωπιών, η μία της ε, ε, αποστολής της Ένωσης, η άλλη του Κοινοβουλίου, ο άλλος από τις αποστολής του Κοινοβουλίου, έφεραν εις πέρας πλήρως τις εντολές τους. Διότι το βασικό ήταν να δούμε ότι δεν υπάρχει καμία ανάμεξη στη, σταθεροποίηση του, στη σταθερότητα τη χώρα και οι δύο αποστολέ κατε, ε, κατεπαιδευματικό τρόπο έφεραν ει πέρα την ε, εντολή του. Πρέπει λοιπόν τέτοιου είδους σταθερότητα να επιζητούμε να υπάρχει παντού χωρίς καμία εξωτερική ανάμειξη. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους συνεργάστηκαν και ιδίως τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου που έκανε εξαιρετική δουλειά για να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας με τη σειρά μας ως παρατηρητές. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Εάν όχι, λίγη η συζήτησή μας σήμερα. Νομίζω κάνατε καλή δουλειά στην αποστολή παρατήρησης ε, στο Λίβανο. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μιας και αυτό ήταν το τελευταίο σημείο για σήμερα, περνάμε απλώς στο 19, διάφορα, δεν βλέπω κανένας να θέλει να θέσει κάτι. Οπότε η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 20 Ιουνίου, 20 και 21 Ιουνίου. Αυτά, σας ευχαριστώ και πάλι για τις εργασίες, για την υπομονή σας. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας από τη Γραμματεία. Κάναμε καλή δουλειά σήμερα. Ευχαριστούμε.